buongiorno a tutti, cominciamo con l'audizione. Σας καλημερίζω. Έχουμε τώρα τον ε, επόμενο υποψήφιο που προτάθηκε από τις Σλοβενικές Αρχές, τον κύριο Μίλαν Μάρτιν Σβίκη. Σβίκλη. Τον καλωσορίζω λοιπόν θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία όπως χθε. Πρόκειται για ένα νέο μέλος, άρα 5 λεπτά για την παρουσίαση, 10 λεπτά στην εισηγήτρια, 20 λεπτά για τις ερωτήσεις των μελών τη Επιτροπή. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για την παρουσίασή σας για 5 λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω στη μητρική μου γλώσσα και να συνεχίσω αγγλικά. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα κυρίως. Πρώτα απ' όλα να σας περιγράψω την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως ειδικό στα δημόσια οικονομικά, ως κεντρικός τραπεζίτης και εργαζόμενος στην Σλοβενία για να διασφαλίσω ότι όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε έναν εξυγχρονισμένο προϋπολογισμό, προετοιμασία δηλαδή και εκτέλεση του προϋπολογισμού και είχαμε τις προϋποθέσεις εκείνες έτσι ώστε και εσωτερικά και εξωτερικά ο έλεγχος ο οποίος γινόταν και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ήταν αποτελεσματικός. Ξεκίνησα εγώ τη αδειοδρομία μου σε κεντρική τράπεζα στη δεκαετία του 80 που τελείωσε βεβαίως με την ανεξαρτησία της Σλοβενίας και τότε είχα αρχίσει να ασχολούμαι με τα δημοσιονομικά ζητήματα δεδομένου του ότι η Ιουκοσλαβία δεν ήταν βιώσιμη όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Στη δεκαετία του 90 εργάστηκα στην Παγκόσμια Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα όσον αφορά τα, τα κράτη-μέλη συνεργαζόταν πάρα πολύ στενά για να διαμορφώσει ένα κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον έτσι ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων να ξοδεύονται σωστά. Επέστρεψα στη Σλοβενία το 1998 και τότε ήμουν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας ε, υπό τον ε, μετέπειτα επίτροπο τον κύριο Ποτότσνικ και φρόντισα στον τομέα των δημοσίων οικονομικών να αποκτήσουμε και νομοθεσία και μια μεθοδολογική βάση που συμπεριλάμβανε και το GFS και το COFOC, την ε, κατάταξη δηλαδή του κράτους, για να καταφέρουμε να γίνουμε κράτος μέλος αποτελεσματικά. Επίσης ήμουν και εθνικός ε, υπεύθυνος για την έγκριση των κονδυλίων ε, των προενταξιακών και καταφέραμε 1η Μαΐου 2004 να γίνουμε κράτος μέλος. Τότε ήμουν υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και φρόντιζα σε όλους τους τομείς ε, που είχαμε επαφή με την Κομισιόν για το κοινοτικό και εκτιμένο να έχουμε την κατάλληλη ε, προετοιμασία. Γιατί είμαι τώρα υποψήφιος ε, για μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Θεωρώ πως υπάρχουν ε, τρία βασικά προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Νομοθεσία με, την, με τις σωστές ε, κατατάξεις κατηγοριοποίησης. Δεύτερον, αποτελεσματικά εθνικά ελεγκτικά όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τρίτον κοινοβουλευτική, κοινοβουλευτικός έλεγχος γιατί έτσι γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το πώς ξοδεύονται τα χρήματα. Και εγώ συνεισέφερα σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία μου στην Σλοβενία σε δύο από αυτά τα τρία σημαντικά στοιχεία. Συνεισέφερα στην ομοθεσία της ε, Σλοβενίας στην, ένα αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που μεταφέρθηκε στην Σλοβενία με το να αντιγράψουμε κάπως σχετικές διατάξεις του Ηνωμένου Βασιλείου και αν με στηρίξετε για να γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσουν πως ε, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα αισθάνονται πως ε, επενδύονται σωστά τα χρήματά τους στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, η έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω Θα ήθελα να σας ε, ε, ρωτήσω το εξής. Έχετε μεγάλη εμπειρία και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο και παρουσιάζεται ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως υποψήφιος. Τώρα όμως, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας, βλέπω ότι έχετε κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες, ε, κυρίως όσον αφορά τη σχέση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού με το Ελεκτικό Συνέδριο που είναι το όργανο στο οποίο προσδοκάτε να συμμετάσχετε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε λίγο περισσότερα σχετικά με τις ιδέες σας αυτές, γιατί εσείς ε, στις ε, απαντήσεις σας ε, αναφέρετε ότι πιστεύετε ότι και τα δύο όργανα έχουν παρόμοιες, παρόμοιες, παρόμοια αποστολή, παρόμοιο σκοπό. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσετε κι εσείς ότι δεν το βλέπετε το θέμα ως μια απλή επικάλυψη, αλλά ως ε, δύο όργανα που έχουν διαφοροποιημένες αποστολές και που η μια συμπληρώνει την άλλη. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Στην έκθεση του κυρίου Μπες, ε, του προηγούμενου προέδρου της Κοκομπού, και ε, στις ομιλίες του ενώπιον του ελεκτικού συνεδρίου τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια ριζική μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Αντί λοιπόν να εκπροσωπούνται τα 27 κράτη-μέλη, να έχουμε ένα όργανο πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό με ε, περιορισμένο αριθμό μελών. Δηλαδή, αντί ε, το σώμα των ελεγκτών να είναι 27 εκπρόσωποι των κρατών μελών, που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο η υπόνοια ότι ο καθή εκπροσωπεί τα συμφέροντα τη ε, χώρα μέλου, να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση με περιορισμένο αριθμό των ελεγκτών, όπου να είμαστε και σίγουροι, αν θέλετε, ότι έχουμε εξασφαλίσει την αμεροληψία και την εξαρτησία του. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώ βλέπετε το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο. Στο ερωτηματολόγιο, στο τέλος, έχουμε την εξής ερώτηση κατά πόσον θα είστε διαδεσμένος να παραιτηθείτε από την υποψηφιότητά σας αν υπάρχει αντιαρνητική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να σας πω ότι η απάντησή σας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ε, καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε την εντύπωση ότι είστε ο καλύτερος υποψήφιος. Μερικές φορές όμως το Κοινοβούλιο ε, ε, ε συμπεριφέρεται με τους δικούς του κανόνες ε, που δεν πολλές φορές είναι οι ίδιοι με τους κανόνες του υποψηφίου. Θα αποσύρετε την αποψηφιότητά σα, λοιπόν εάν το Κοινοβούλιο θεωρήσει ότι δεν είστε ο ιδεώδης υποψήφιος. Βεβαίως αυτό δεν, δεν προδικάζω το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Απλά και μόνο σας ρωτώ στην περίπτωση που. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ναι, πιστεύω ότι η Κοκομπού ε, και, το Ευρωπαϊκό ε, ε, ε, Ελεκτικό Συνέδριο έχουν παρόμοια αποστολή. Θα έλεγα ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο, με την εξή έννοια. Όταν η Κοκομπού προβαίνει σε ε, εξέταση μια συγκεκριμένη έκθεση και κάνει μια έκθεση, αυτή η έκθεση έχει να κάνει με το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλέ φορέ και τα, ε, και τα κρατημέλη ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Εμεί έχουμε παρόμοια κατάσταση και στη Σλοβενία. Παλιά γινόταν ακροάσεις όπου τα μέλη του Κοινοβουλίου υπέβαλαν ερωτήσεις στα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. που θα υποβληθούν συνέχεια στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ε, ακριβώς το ένα όργανο συμπληρώνει το άλλο. Με την έννοια ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου εργάζονται για εσά κατά κάποιο τρόπο. Και εσείς αξιοποιείτε τα ευρήματα του Ελεκτικού Συνεδρίου για να μπορέσετε να υποβάλλετε ερωτήσεις και βεβαίω με βάση τα δικά μα τα ευρήματα, τα ευρήματα του Ελληνικού Συνεδρίου, να προβείτε σε αλλαγέ στην νομοθεσία, σε αλλαγέ στι διαδικασίε. Έτσι ώστε να έχουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση και χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων. Εάν βρούμε λοιπόν ένα modus operandi όπου τα μέλη του Ελευθερικού Συνεδρίου και οι σχετικέ εκθέσει αποτελούν τη βάση για τη δική σα εργασία, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα βήμα προ τα εμπρό. Και βέβαια αυτό το θέμα συνδέεται ιδιαίτερα με το θέμα τη δική μου παρέτηση, εάν δεν γνωμοδοτήσετε θετικά. Κοιτάξτε, ήρθε εδώ για να παρουσιάσω τον εαυτό μου και πιστεύω, ακριβώ γι' αυτό είμαι υποψήφιο, πιστεύω ότι με βάση την επαγγελματική μου εμπειρία δεν υπάρχει κανένας μείζον λόγος για τον οποίο να μην μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Έτσι ώστε και εγώ με τον ρόλο μου και τις αρμοδιότητές μου να σας βοηθήσω και να και να συμβάλλω προς την αξιολόγηση ε, της, της, της χρησιμοποίησης των χρημάτων των, των φορολογουμένων. Πιστεύω ότι έχω την απαραίτητη εμπειρία και από τη χώρα μου, έτσι ώστε ε, να συμβάλλω προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ε, αποτελεσματικής δημοσιονομικής εποπτείας με στόχο την χρηστή διαχείριση και τη δημιουργία μιας νοοτροπίας χρηστής διαχείρισης. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια αυτά και με βάση αυτά που σας είπα, αν δεν έχω την εμπιστοσύνη σας, θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να συνεργαστώ μαζί σας. Γι' αυτό ε, υπολογίζω στη δική σας υποστήριξη. Και όσον αφορά την επόμενη ερώτηση, κατά πόσο δηλαδή το σώμα των ελεκτών θα πρέπει να αποτελείται από 27 μέλη, όχι η, θεωρία οργάνωση λέει ότι όταν έχουμε πάνω από 7 ανθρώπου σε ένα δωμάτιο, είναι δύσκολο να γίνει συζήτηση. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Η ιδέα λοιπόν των τεσσάρων σωμάτων όπου ένα, ένας περιορισμένος αριθμός μελών θα προβαίνει σε προακροάσεις ε, ε, των επιμέρους εκθέσεων πριν συζητηθεί στην Ολομέλεια των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου, ίσως αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αλλά βεβαίως δεν έχω, κατέχω όλες τι πληροφορίες αυτή τη στιγμή ώστε να κάνω, ε, να τοποθετηθώ οριστικά. Αλλά έχω την άποψη ότι εάν η εργασία οργανωθεί με ένα τέτοιο τρόπο, που ε, μια μικρότερη ομάδα των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου προετοιμάζει τις εκθέσεις και τις συζητά σε ένα είδος προκαταρκτικής ακρόασης, και δίνει τελικά τι οριστικέ πληροφορίε ε, στην Ολομέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, τότε θα έχουμε αυξήσει και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου θα βοηθήσει και το Ελεκτικό Συνέδριο και τα μέλη για να μπορέσουν να εργαστούν προς το βέλτιστο συμφέρον της Κοκομπού αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν εσείς ε, εξετάζετε ε, και επιβλέπετε το πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Κοιτάξτε. Με βάση τη μακρά σας εμπειρία, είχατε σημαντική σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα πρέπει να γνωρίζετε γιατί ε, βεβαίω οι υποψήφοι προετοιμαστήκατε πολύ καλά, ότι μία από τι πτυχέ όπου ε, συναντάμε συχνά προβλήματα στην Επιτροπή μα ε, είναι το θέμα του ελέγχου τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που συμμετέχει σε προγράμματα συνεργασίας με άλλα ε, διεθνή ιδρύματα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, με άλλους διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις δικές σας ιδέες και πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς στο να ασκήσουμε πιο αποτελεσματικά τον έλεγχο αυτό. Και τέλος, μου προξένησε έκπληξη το γεγονός ότι όταν σα ρώτησα, αν θέλετε να μου το διευκρινίσετε, να το ξεκαθαρίσετε. Στην ερώτηση αν έχετε προβλήματα με τη δικαιοσύνη, μιλήσατε για το διαζύγιό σας. Κοιτάξτε, ε, δεν πρέπει να είμαστε μόνο ε, τίμοι, αλλά και να φαινόμαστε έτσι. Να, μας, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι δεν, δεν υπάρχει καμία ανάμειξη της ιδιωτικής σας ε, ζωής ε, ε, με την μελλοντική άσκηση των καθηκόντων σας ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. On the question of effectiveness of σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διεθνών χρηματοδοτικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προσπαθειών τις οποίες κάνει στα πλαίσια της βοήθειας για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω 6-7 χρόνια εμπειρία στην Παγκόσμια, στην Παγκόσμια Τράπεζα και υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα χρηματοδοτικά όργανα και στους άλλους οργανισμούς που κινούνται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών. Ένα παράδειγμα. Εγώ σαν οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας πήρα μέρος στη διατύπωση του προγράμματος ανοικοδόμησης της Βοσνίας Ευζεγοβίνης. Συνεργαστήκαμε και με τα ευρωπαϊκά όργανα και υπήρξαν κάποια προβλήματα με ορισμένα άλλα όργανα επίσης διεθνή. Όταν λοιπόν δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όταν υπάρχουν πολλαπλής, πολλαπλή διεθνείς οργανισμοί, είναι σημαντικό κάποιος να έχει μια ηγετική ε, θέση. Η Παγκόσμια Τράπεζα στη Βοσνία Ευζεγοβίνη, στην ανοικοδόμησή της, ήταν θα έλεγα ηγέτης. Συνεργαστήκαμε και με τα υπόλοιπα διεθνή οικονομικά όργανα και πήραμε νομίζω τα κατάλληλα μέτρα. Κάποιες από τις εμπειρίες που βιώσαμε θα μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω και σε αυτά τα οποία σκοπεύω να κάνω στο μέλλον. αλλά δεν θα ήθελα να πω δημόσια ότι ό,τι γίνεται σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι επιτυχές όταν τα χρήματα δίδονται, δανείζονται, μπας περιπτώσει, υποτύπων δανείου ε, και σκοπεύει το χρηματοδοτικό όργανο τα οποία τα χορηγεί να τα ανακτήσει σε κάποια φάση, αυτό ίσως είναι μερικές φορές καλύτερο από το να δίδονται υπό τη μορφή δωρεάς. Τώρα σχετικά με το διαζύγιο. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες γύρω από το διαζύγιο μου στη χώρα μου και πράγματι υπήρξαν κάποιοι υπεύθυνοι της ε, δημόσιας διοίκησης που θεώρησαν ότι ήμουν πάρα πολύ σκληρό σε σχέση με την πράσπιση των συμφερόντων μου. Αλλά η διαδικασία είναι ανοιχτή και τρέχουσα. Η κυρία Αντρεάσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Σβίγκελ. Βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας ότι από το 2004 μέχρι το 2008 ήσασταν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Δημοσιονομικό Έλεγχο. Ήσασταν υπεύθυνο για ένα πρόγραμμα συνεργασίας με το ελεγκτικό συνέδριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί αποφασίσατε να συνεργαστείτε με τους Βρετανούς και όχι με το ε, ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών. Δεύτερη ερώτηση. Αν μπείτε στη θέση του Ευρωπαίου φορολογούμενου, πιστεύετε ότι η DAS, η δήλωση αξιοπιστίας για το 2008, πρέπει να ικανοποιεί έστω κατελάχιστον τον Ευρωπαίο φορολογούμενο για τη σωστή χρήση των χρημάτων. γιατί συνεργαστήκαμε με τους Βρετανούς. Το κάναμε αυτό στα πλαίσια της δυνατότητας που μας παρήχε το ε, λεγόμενο μεταβατικό μέσο για την ένταξη. Μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα ελεγκτικά συστήματα των ε, κρατών μελών. Είχαμε προσφορές από τρεις χώρες, και ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τους Βρετανούς ήταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς τους, το κόστος και η ικανότητα του ελεγκτικού συνεδρίου του Ηνωμένου Βασιλείου να μας παρέχει άμεσα περιεχόμενο και πληροφορίες, έτσι ώστε η αντίστοιχη επιτροπή του Σλοβενικού Κοινοβουλίου του οποίου ήμουν πρόεδρος να συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών της Κάτω Βουλής. Υπήρξε η δυνατότητα ανταλλαγής επισκέψεων. Παρακολουθούσαμε συστηματικά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη σελίδα 12, τελευταία παράγραφος και στη σελίδα 16, στη δεύτερη παράγραφο, υπάρχει ένα λάθος λέγοντας ότι το PAC είναι η Επιτροπή Πολιτικής Δράσης, ενώ δεν είναι έτσι, είναι η Επιτροπή ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου. Εν πάση περιπτώσει ε, πήραμε πολλές εμπειρίες, θετικές εμπειρίες και στο τέλος υιοθετήσαμε ένα νέο κανονισμό λειτουργίας της Αρμόδιας Επιτροπής στη Σλοβενία που έδινε τη δυνατότητα στα μέλη αυτής της Επιτροπής να λειτουργήσουν διακομματικά να μην παίξουν τον ρόλο τους σαν δεξιοί ή σαν αριστεροί, αλλά να μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στους αξιωματούχους της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες να βασίζονται στις γνώμες και στις απόψεις τις οποίες είχε συλλέξει το Σλοβενικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή ήταν μια πολύ καλή πρακτική την οποία κερδίσαμε και είναι και, και η απόδειξη του συμπληρωματικού ρόλου τον οποίο παίζουμε. Τώρα το 2008 και για τη δήλωση αξιοπιστίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει η κοκομπή και η κομπού. Δεν θα ήθελα εδώ να, ε, πω, να ισχυριστώ ότι η μεθοδολογία και η δεδομένη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο κινδύνου και στο ύψος ε, του ελέγχου παρέχουν τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας τα οποία θα ικανοποιούσαν το ελεγκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει θετικά. Βασικός ρόλος κάθε ελεγκτικού οργάνου όπως και του ευρωπαϊκού είναι να επιδιώκει τις ε, ε, αλλαγές προς το καλύτερο. Και εδώ έρχεται και ο δικός σας ρόλος, ρόλος ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που δείχνει ότι τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο φέρει εις πέρας τον δημοσιονομικό έλεγχο και προστατεύει τα συμφέροντα των φορολογουμένων. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προσπάθειες αλλαγής της μεθοδολογίας και οι προσπάθειες περαιτέρω εμβάθυνσης της ποιότητας των ενδιαμέσων μορφών ελέγχου και των ενδιαμέσων εκθέσεων είναι κάτι το οποίο θα προσφέρει πολλά στην ποιότητα των εργασιών σας. Ο κύριος Ντόιτς. Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Δυστυχώς δεν λάβαμε πληροφορίες τις απαντήσεις δηλαδή στο ερωτηματολόγιο. Αλλά έχουμε τις ε, πληροφορίες από το 2004. Είναι γνωστό πως τότε το Σλοβενικό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε την υποψηφιότητά σας για την Προεδρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ε, Σλοβενίας τα κόμματα της αριστεράς είχαν την ε, πλειοψηφία τότε στο κοινοβούλιο οπότε δεν νομίζω να ήταν πολιτικό το ζήτημα κάτι άλλο θα ήταν εάν η Βουλή της Σλοβενίας δεν σας θεωρήσε ικανό να γίνεται. Πρόεδρο του Ανεκτικού Συνεδρίου τη Χώρα σα πώς ε, να σας θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ικανό για να γίνετε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου. Δεύτερον, η Αγέλα Σέντερ ανέφερε ήδη το εξή. Κάτι πολύ απλό. Η... Εάν η Επιτροπή μας δεν υποστηρίξει την υποψηφιότητα κάποιου, τι θα γίνει, θα, θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας. Ε, απλό είναι, μία απλή απάντηση με ναι ή όχι. Αν δεν θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας, ε, εντάξει, δεκτών. Αλλά νομίζω ότι δεν απαντήσατε. Με απλά λόγια σε αυτή την ερώτηση. Θέλω απλά ένα ναι ή ένα όχι από εσάς. Και τα δύο δεκτά. Απλά θα θέλαμε να ξέρουμε εάν είστε διατεθειμένος να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν δεν σας προστηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο ερωτήσεις. Πράγματι το τέλος του 2003 ήμουν υποψήφιος για πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου στην Σλοβενία. Με βάση τη δουλειά μου το 99 και 2000, όταν εισήχθη διαφανής θα έλεγα νομοθεσία, έγινα γνωστός στην Σλοβενία ως κάποιος ο οποίος είναι ανεξάρτητος, αλλά ταυτόχρονα και κάποιος ο οποίος είναι δύσκολος να μεταπιστεί, αν θεωρεί πως ε, κάτι είναι σωστό. Πράγματι ήμουν υφυπουργό τη κυβέρνηση και φανταζόταν κανεί πω ε, η Αριστερή πλειοψηφία θα με υποστήριζε ω ε, πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου. Γιατί δεν το έκαναν δεν ξέρω. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και χρειαζόταν βεβαίως η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Και οι φήμες βεβαίως έλεγαν ε, πως ε, δεν ε, θα μπορούσα να χειραγωγηθώ εύκολα. Οπότε λέγανε το να δώσουμε σε αυτό το άτομο μία εντολή 9 ετή ειδικά όταν θεωρούσαν ότι θα κέρδιζαν τις εκλογές ε, του χρόνου, θεώρησαν καλό να μην μου δώσουν την εντολή. Η ίδια κυβέρνηση μετά μου ζήτησε να αντικαταστήσουν τον κύριο Ποτότσνικ ως ε, υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων λόγω έτσι, ως, ως τεχνοκράτης ε, που είχα ασχοληθεί με ζητήματα σημαντικά για την Σλοβενία. Οπότε δεν θα έλεγα πως ε, δεν έρχα της ε, εμπιστοσύνης του Σλοβενικού Κοινοβουλίου γιατί όταν δεν ήταν μυστική ψηφοφορία με υπερψήφισαν για τρεις του Υπουργού. Αλλά στη μυστική ψηφοφορία πράγματι με απέρριψαν. Τα δε κεντροδεξιά κόμματα το 2008 με απέρριψαν, εντάξει εκεί ήταν πολιτικό το ζήτημα. Και πράγματι είπα ε, και στην απάντησή μου πως είμαι ε, ανεξάρτητος εδώ πέρα. Δεν μπορώ τώρα να σας πω ναι ή όχι. Θα έρθω εδώ πέρα, θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι στην 20 η μου σταδιοδρομία ε, είμαι τεχνοκράτης. Εάν δεν επαρκεί αυτό για τη στήριξή σας, ε, είναι πολύ δύσκολο να... να εργαστώ και ως ε, μέλος χωρίς ε, τη στήριξή σας. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι προφανής. Αν δεν με στηρίξετε θα γυρίσω στο σπίτι μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε τον υποψήφιο. Ε, από την Σλοβενία και τώρα περνάμε στις ακροάσεις ε, ε, που αφορούν την επιβεβαίωση υποψηφίων. Εδώ έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε 20 λεπτά για κάθε υποψήφιο και ξεκινάμε με τον υποψήφιο που προτάθηκε από τις Εθνικές Αρχές, τον Γιάνν Κίνστ. Α, παρουσίαση και των τριών. Κίνστ, Κάλτζουλάιντ και Lundborgs. Ε, αντίστοιχα από τι εστονικέ και λετονικές αρχές. Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, η διαδικασία είναι γνωστή. Τα μέλη εδώ που έχω δίπλα μου είναι γνωστά ε, στα μέλη της Επιτροπής μας. Θα πρέπει ο καθένας από τους τρεις υποψηφίους να κάνει μια πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση και να δώσω αμέσως μετά το λόγο στην Αγιάλα Σέντερ. Κύριε Κίνστ, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και ζητώ την εμπιστοσύνη σας για μια δεύτερη εντολή. Όπως γνωρίζετε, εγώ πήγα στο ελεγκτικό συνέδριο 6 χρόνια, πριν 6 χρόνια και ανέλαβα τις εξωτερικές δράσεις τις οποίες προσπάθησα να εργαστώ μέχρι τώρα Κατά τη διάρκεια της εντολής μου δύο φορές χρήστηκα υπεύθυνο για την ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και για τον τομέα των εκθέσεων ελέγχου επιδόσεων στον τομέα πάντα της βοήθειας για την ανάπτυξη. Είχα τη δυνατότητα να είμαι εδώ στο παρελθόν και να σας υποβάλω τρεις ειδικέ εκθέσεις και χαίρομαι γιατί και οι τρεις αυτές εκθέσεις έγιναν θετικά δεκτές η ειδική έκθεση για το περιβάλλον, για τον τομέα της υγείας και για τη διαχείριση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στο ελεγκτικό συνεδρίο ασχολήθηκα και με οριζόντια θέματα όπως τα θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και πάντα είμαι υπεύθυνο για τον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Ασχολήθηκα και μεθοδολογικά θέματα στον τομέα της ε, διαδικασίας ελέγχου για την άμεση δημοσιονομική βοήθεια. Αυτά συνοπτικά είναι αυτά τα οποία έκανα τα τελευταία χρόνια. Είχα την τιμή να συνεργαστώ επανειλημμένα μαζί σας και θα ήθελα να μου ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας για μια ακόμη περίοδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Καλεουλάιτ από την Εστονία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε την δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κοκομπή μετά από έξι χρόνια που ήμουν υπεύθυνη για ορισμένα θέματα στο ελεγκτικό συνέδριο. ξεκίνησα σαν το μέλος, το υπεύθυνο του Συνεδρίου για τις Εσωτερικές Πολιτικές και της Έρευνας και τώρα είμαι υπεύθυνη για την αξιολόγηση επιδόσεων στον τομέα της συνοχής. Όπως και οι συναδελφοί μου έχω πάρει μέρος στην Επιτροπή ε, Διαχειριστικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προέδρευσα της ε, Επιτροπής αυτής για δύο χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα θέματα πληροφορικής. Έχω, κάνει, έχω συντάξει την έκθεση την ειδική για το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Έχω λάβει την δική σας υποστήριξη για όλες τις ειδικέ εκθέσεις τις οποίες έχω πάρει μέρος, όπως επίσης και για τις συζητήσεις τις οποίες έχουμε κάνει μεταξύ μας. Ήμουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ελληνικής Επιτροπής και πρόεδρος της για ένα από τα τρία χρόνια και ήμουν και στην ε, ομάδα αυτοαξιολόγησης του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ε, εμπειρία μου όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας ε, σε ένα think tank που εξετάζει το μέλλον των δηλώσεων αυτών αξιοπιστίας ε, για τις οποίες βέβαια και η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη. Αναμένω λοιπόν τις ερωτήσεις σας και ελπίζω να με εμπιστευτείτε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Ίγκορ Σλουτμπορξ, τον υποψήφιο πρωτάθλημα της Λιτωνικής Αρχές. Uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι εδώ μαζί σας και να παρουσιάσω το τι έκανα τα πρώτα έξι χρόνια της εντολής μου. Πρώτα απ' όλα ήμουν το μέλος υπεύθυνο για τον τραπεζικό δανεισμό και με αυτή την εντολή ήμουν υπεύθυνο για, το για τα κεφάλαια 10 και 11 στην ετήσια έκθεση του συνεδρίου. Επίσης συνέταξα και μια γνωμοδότηση του συνεδρίου και πρόσφατα παρουσίασα δύο ειδικέ εκθέσεις Συμβουλευτική Επιτροπή, μία για την στρατηγική διαχείριση της Κομισιόν και μία δεύτερη για τα τραπεζικά μέτρα που αφορούν τα προγράμματα ΜΕΝΤΑ. Όσον αφορά τα οριζόντια καθήκοντα, από το 2006 ήμουν μέλος Διοικητικής Επιτροπής και από το 2008 προεδρεύω στην Διοικητική αυτή Επιτροπή του Συνεδρίου. Και οι τρεις ε, εδώ συνάδελφοι είμαστε, είμαστε μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και η συνάδελφος ε, η κυρία Καλιουλάιντ προηγήθηκε ως πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνο για μια ειδική έκθεση που θα ασχοληθεί με το πολύ σημαντικό ζήτημα της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ήμουν και μέλος μιας ομάδας εργασίας που ασχολείται με τα ζητήματα της τρέχουσας οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Αναμένω την στήριξή σας λοιπόν για μια δεύτερη θητεία και ελπίζω να με εμπιστευτείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τώρα να Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ για να υποβάλει τυχόν ερωτήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Σε αυτή τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των υποψηφίων, υποψηφίων που γνωρίζουμε πολύ καλά και μέσα από την δράση τους και την συνεργασία τους με την Επιτροπή, θα επικεντρώσω την προσοχή μου στο μέλλον. Δεδομένης της ε, μεταρρύθμισης στο ελεκτικό συνέδριο, ε, να εξελίξει και, της, ε, και του νέου σταδίου, της νέας φάσης που ε, μας κάνει να ελπίζουμε ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Κίστε, να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Κοιτάξτε, η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, δεν ε, χρησιμοποιεί μόνο από λειτουργική άποψη τις δικές της ακροάσεις, αλλά ζητάμε περισσότερα για να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι εντοπίζονται. Με αυτή την έννοια, όσον αφορά την εξωτερική δράση, εντοπίσαμε ένα πρόβλημα σημαντικό με, τις διεθνείς, με διεθνείς οργανισμούς. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πώ ε, πώς θα μπορούσαμε στο μέλλον να βελτιώσουμε σημαντικά αυτή την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εδώ αναφέρεται η ανάγκη κεντρικού σχεδιασμού για τον καλύτερο έλεγχο, δηλαδή να μειωθούν ε, οι τομείς εξωτερικής δράσης, να μειωθεί ο ρυθμός και η διάχυση ανάμεσα στις μη κυβερνητικέ οργανώσει. Άρα, ο κίνδυνος ποιος είναι, να μην φτάσουμε τελικά στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που βρίσκονται επί τόπου. Όσον αφορά λοιπόν την εξωτερική δράση και τη οποία ε, το διπλωματικό τμήμα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο τι θα γίνει με αυτέ τι οργανώσει που δρούν επί τόπου και που είναι πάρα πολύ σημαντικέ ε, και για την προώθηση τη δράση, την προβολή τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνο να τι χάσουμε από, το, ε, από τα μάτια μα στο μέλλον και να μην μπορούμε πλέον να αξιοποιήσουμε τη δική του ικανότητα. Να συνεχίσω. Μάλιστα. Στην κυρία Καλβιλάιτ, θα ήθελα να σα πω ότι Ε, ορισμένοι ε, ε, ε συνάδελφοι και συντροφοί μου μου έλεγαν ότι καλύτερα θα πρέπει να σας συγχαρούμε παρά να σας κάνουμε ερωτήσεις. Αλλά ε, θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά την, την ομάδα peer review, την αυτοαξιολόγηση, θα ήθελα να μας πείτε το εξής. Τώρα που μόλις εγκρίθηκε η μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου, αυτό το τμήμα ε, του ελέγχου του ελεγκτή που μας προσφέρει εγγύησεις. Πού πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να βρίσκονται οι βάσεις, πού θα πρέπει να βρίσκονται τα βασικά στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μιλώ για τον έλεγχο του, του ελεγκτή. Και όσον αφορά τις δηλώσεις αξιοπιστίας DAS, να σας ρωτήσω το εξής, το οποίο προέκυψε και μέσα από τις πρόσφατες συζητήσεις όσον αφορά τα οικονομικά έτη, τα οποία δεν, ε, ε, ε, μάλλον τε, τε, τις οικονομικές περιόδους που δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο έτος, αλλά γενιές αν θέλετε, χρονολογικές. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, αυτό που βλέπει τελικά ο πολίτη, να μην είναι μόνο η χρονιά που είχε καταστροφικά αποτελέσματα, αλλά ολόκληρο τον κύκλο με τα προβλήματα και με, τις, και με τα σημεία στα οποία δεν υπήρχαν, τα παρατυπίε, τα προβλήματα. Και τέλο, όσον αφορά τον κύριο Λούτσπορτ, να σα πω το εξή. Να σα ρωτήσω το εξή. Τόσο στην Επιτροπή Διοικητικών Υποθέσεων που μα απασχολεί βεβαίω όταν ε, έχουμε να εξετάσουμε την απαλλαγή του ηλεκτρικού συνεδρίου. Εδώ θα ήθελα να μου πείτε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και πώ θα προωθήσετε τη βελτίωση τη οργάνωση αλλά και τη αποτελεσματικότητα του ηλεκτρικού συνεδρίου προ την κατεύθυνση αυτή. Και δεύτερον, σε σχέση με την οικονομική κρίση, μία από τι πτυχέ που τα κράτη-μέλη αλλά και όλοι οι θεσμοί ε, απασχόλησε δηλαδή ε, όλους τους θεσμούς, είναι ακριβώς η απλοποίηση. Ε, πρέπει λοιπόν να διευκολυνθούν οι διαδικασίες όσον αφορά τα προγράμματα και τις, ε, ε τα ευρωπαϊκά προγράμματα της ευρωπαϊκής δράσης. Αυτό βεβαίως να μην γίνεται εις βάρος του δημοσιονομικού ελέγχου, δηλαδή αποτελεσματικότητας ε, και εγγυήσεων ε, της σωστής δαπάνης των χρημάτων. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική 2020 και εκεί θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να μάθω και τη δική σας άποψη του ζητήματος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κίνστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στο ζήτημα των διεθνών οργανισμών Πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοχετεύει πολλά λεφτά μέσω διεθνών οργανισμών σε περιπτώσεις τις οποίες ε, οι οργανισμοί αυτοί όπως είναι ο ΙΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα είναι εδρεωμένοι σε κάποιες χώρες ε, που βγαίνουν από μια κρίση ανθρωπιστική κτλ γνωρίζετε πως πρόσφατα δημοσιεύσαμε τον έλεγχο που λέγεται ΟΗΕ 1 όπου αξιολογούμε αν η Κομισιόν ε, έχει αποφασίσει σωστά να διοχετεύσει χρήματα μέσω διεθνών οργανισμών και συγκρίνουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου και ήμασταν αρκετά επικριτικοί ως προς αυτό σε αρκετές ε, περιπτώσεις. Μας φάνηκε ως μια διέξοδος ε, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ισχύει τώρα όσον αφορά την προετοιμασία του δημοσιονομικού κανονισμού γνωρίζετε πως υπάρχει η δυνατότητα ή προτείνεται η δυνατότητα πως ε, η Κομισιόν θα πρέπει να διαχειρίζεται αυτά τα καταπιστεύματα πολλαπλών δωρητών και αυτό νομίζω, πολλών δωρητών. Αυτό νομίζω είναι θετικό ειδικά, καθώς η Κομισιόν είναι μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής και αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Η πιο σκανδαλώδης περίπτωση το ήταν το ταμείο για το κλείσιμο του, του Τσερνομπίλ όπου έδωσε χρήματα χωρίς να έχει λόγο η Κομισιόν. Βεβαίω τα ζητήματα των διεθνών οργανισμών είναι ευαίσθητα και ίσως ε, θα ξέρετε πως ε, ένα άλλο κίνητρο για την διαχείριση από την ίδια την Κομισιόν είναι η πρόσβαση στα έγγραφα και για την Κομισιόν και για το ελεγκτικό συνέδριο και για την επιβολή της σωστή λειτουργία της συμφωνίας ε, που επιτρέπει στην Κομισιόν και στο συνέδριο να ελέγχει τα έγγραφα όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ξέρετε πως υποβάλαμε μακροσκελής ε, ε, ελέγχους όσον αφορά δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα πώς η Κομισιόν εμπλέκει τις ΜΚΟ ως εταίρους για τις στρατηγικές αποφάσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία Αναφέρεται αυτό στο Κομισιόν σε πολλά πολιτικά όγγραφα, αλλά εμείς ήμασταν επικριτικοί, γιατί είναι μεγάλη η αλλαγή, αλλά δεν έγινε αυτό επί τόπου. Δεύτερον, ήμασταν λιγότερο επικριτικοί όσον αφορά την διαχείριση της, ε, των ΜΚΟ ως ε, των φορέων εκείνων που θα εφάρμοζαν τα προγράμματα της Κομισιόν π.χ. για την απόκτηση διοικητικής κανότας και τα λοιπά κατάρτισης. Επειδή αναφέρατε το EIS, επειδή ξέρετε πως αυτό το ζήτημα ακόμα εκρεμεί και θα εκρεμεί στο μέλλον, ελπίζω να μην επηρεάσει την προσέγγιση αυτή της Κομισιόν προς τους ΜΚΟ ως έτσι, χειραφετημένων εταίρων στην αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί είχα την δυνατότητα να πάω σε μέρη που εργάζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πραγματικά υπάρχει πολιτική αστάθεια σε αυτές τις χώρες και είναι μία από τις λίγες εγγυήσεις ε, της συνέχειας της βοήθειας. Οπότε, από όσο ξέρω, οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται, αλλά υπάρχει αυτό το οποίο διάβασα είναι πως η Κομισιόν θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τα συγκεκριμένα αυτά προγράμματα και την εφαρμογή της βοήθειας και ελπίζω να μην βλάψουμε την διαδικασία αυτή της εμπλοκής των ΜΚΟ στην αναπτυξιακή συνεργασία. Η κυρία Καλιουλάιντ. Ευχαριστώ και από τα peer review και από την αυτή χρειάστηκε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και γι' αυτό ε, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το θέμα των επιμέρους σωμάτων στο εσωτερικό του ελεγκτικού συνεδρίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των διαδικασιών επικοινωνίας και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Ένας ελεγκτής είναι αξιόπιστος μόνο εφόσον είναι διαφανής και η διαφάνεια ε, εντάσσεται, έγκυται μάλλον και στο θέμα της διαδραστικής σχέσης και με την Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη. και θα πρέπει εμείς να ε, μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τα κράτη-μέλη σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μειώσουμε τα ποσοστά λάθους των στοιχείων επικοινωνίας τα οποία λαμβάνουμε ε, από τα κράτη-μέλη. Αυτά ε, ε, τα λάθη προέρχονται κυρίως από τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται και επηρεάζουν αρνητικά τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τη σύνθεσή του. Φυσικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από όλου να εφαρμόσουν τη δική μας μεθοδολογία, αλλά αν η δική μας μεθοδολογία είναι διαφανής, δίκαιη και αποτελεσματική, νομίζω ότι και άλλοι θα μας ακολουθήσουν και αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά σε επίπεδο ποιότητα την οποία μπορεί να δώσει το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, σε σχέση με την πολιετή βάση και πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι επιλύονται τα προβλήματα στον τομέα της συνοχής. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, δεν είμαι βεβαία ότι πράγματι έχουν επιληθεί τα περισσότερα προβλήματα. Η έκθεση για το 2008, ακόμα και στις δαπάνες αντικατάστασης, έγιναν πάρα πολλά λάθη και ε, ιδιαίτερα στο κλείσιμο των προγραμμάτων και στην προετοιμασία του κλεισίματος των προγραμμάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο εκ των υστέρων μόνο παραμένει αυτό το οποίο βλέπει τι παραμένει ε, σε εκκρεμότητα μετά από το κλείσιμο των προγραμμάτων. Σχετικά με τις αλλαγές γύρω από τα νέα προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι έχει σεβαστεί μέχρι τώρα τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με ε, τις καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν και άρχισαν επιτέλους οι πληρωμές. Και φαίνεται ότι οι πρώτες πληρωμές περιλαμβάνουν πολύ λιγότερα λάθη από ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί οι πρώτες πληρωμές να γίνονται με σωστό τρόπο αλλά το τι θα ακολουθήσει δεν έχουμε εγγυήσει για το αν θα περιλαμβάνουν περισσότερα λάθη ή όχι. Για να πείσουμε το κοινό λοιπόν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, να δείξουμε τι σημαίνει έλεγχος, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνουν τα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι το να σηκώνουμε, να κραδένουμε ακόμα αν θέλετε την σημαία την κοινοτική στις τριμερείς συναντήσεις είναι κάτι το θετικό σε επίπεδο επιχειρημάτων. Δεν θα πρέπει φυσικά να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στα λάθη τα οποία έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και ποια είναι συνολικά τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στον τομέα της συνοχής και έτσι θα καταλάβουμε αν για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές ο τομέας της συνοχής θα πρέπει να παραμένει ως έχει ή να αλλάξει τα προβλήματα τα οποία εμπεριέχονται αν θέλετε είναι ενδογενή στο σύστημα μικτής διαχείρισης είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την μελλοντική εργασία της, της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων, θα ήθελα να πω ότι όπως αναφέρθηκε και στη στρατηγική του ελεκτικού συνεδρίου για το 2009-2012, έχουμε τους εξής στόχους. Ε, μεγιστοποίηση της, ε, ε, ε, του αντικτύπου και βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων. Και αυτό συνδέεται και με το, και με το εξής στα πλαίσια της ε, Διοικητικής Επιτροπής πρέπει ε, να καταρτιστούν, πρέπει να καταρτιστεί μία σειρά από πολιτικές ευρέως φάσματος ε, στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, των ανθρωπίνων πόρων και να αναφερθώ σε αυτό το τελευταίο. Πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι για τη βελτιστοποίηση των κινήτρων του προσωπικού. Και μία άλλη σημαντική πτυχή έχει να κάνει με την κινητικότητα του προσωπικού. Να υπάρξει δηλαδή μια κάποια επιτροπή, περιτροπή και εναλλαγή ε, των ελεγκτών που να ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο τομέα και μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 6-8 ετών και βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαίτερε περιπτώσει να, να, μετατίθενται σε άλλου τομεί έρευνα και ελέγχου. Να προσθέσω επίση και το εξή. Όπω τα γνωρίζετε ενδεχομένω, το Συμβούλιο των Υπουργών πρόσφατα ενέκρινε ε, τους, ε, το νέο καταστατικό, τον νέο ιστορικό του συνεδρίου. Και ε, εμείς ε, εργαζόμαστε σκληρά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των κανόνων αυτών. Θα, υπάρξει, θα υπάρξουν εξή ε, αλλαγές. Θα υπάρξει αυτή η εργασία στα, στους, επιμέρους σώματα και θα το δούμε αυτό από το τέλος του θέρους κτλ. Αλλά ως αντιστάθμισμα θα έχουμε την ενισχυμένη Διοικητική Επιτροπή. Ενισχυμένη με την έννοια ότι ο πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου θα είναι και πρόεδρος αυτή τη συγκεκριμένη επιτροπή τη διοικητική επιτροπή. Και οι πρόεδροι των επιμέρου σωμάτων θα είναι μέλη τη διοικητική επιτροπή. Τέλο, να σα πω το εξή. Το ελεκτικό συνεδρίο είναι ένα οργανισμό που όλο και αυξάνεται η δράση του και βεβαίω πρέπει να δούμε το ζήτημα των πόρων πριν από ορισμένα χρόνια εντοπίστηκε το ζήτημα αυτό όταν είχαμε έλλειψη ελεκτών. Είχαμε 56 θέσεις ελεκτικές και με τη δική σας τη βοήθεια ε, καλύψαμε τις 32. Πράγμα το οποίο σημαίνει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε άλλους 24 ε, ανακοινώθηκε από τι ε, δημοσιονομικέ αρχέ ότι λαμβάνοντα υπόψη την οικονομική κρίση δεν είναι πιθανό να καλυφθούν αυτέ τι θέσει. Και αυτό είναι κατανοητό. Άρα προσπαθούμε να δούμε πώ θα μπορέσουμε να μεταθέσουμε προσωπικό από, ε, ε, ε, από άλλα καθήκοντα στον τομέα του ελέγχου. Έτσι ώστε να αυξήσουμε του ελεγκτέ σε εσωτερικό επίπεδο. Με εσωτερικέ μεταθέσει. Όσον αφορά τις βελτιώσεις ε, εν ώψη και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχει μια ομάδα εργασίας μέσα στο συνέδριο και εγώ είμαι ένα από τα τρία μέλη της Επιτροπής αυτής και προσπαθούμε να εξετάσουμε διάφορα ζητήματα. Και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ενδεικτικά το, το πρόγραμμα ανάκαμψη ευρωπαϊκή οικονομία, όπου προβλέπεται, περισσότερα ταπάνε σε, σε ορισμένου τομεί και ε, περισσότερε προκαταβολέ σε, σε άλλου. Αυτό βεβαίω ενέχει συμπληρωματικού κινδύνου και το αναγνωρίζω. Διότι ακριβώ αυτή η τομή είναι και η προβληματική. Εξακολουθούμε επίση να εξετάζουμε την υποστήριξη του συζυγίου πληρωμών που ε, αυτή τη στιγμή αφορά, ε, διευρύνθηκε προ τρία κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη Λετωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Στην έκθεση του 2008 αναφερθήκαμε σε, ορισμένες, ε, ε, σε ορισμένα στοιχεία και τώρα εξετάζουμε και την περίπτωση να προβούμε σε έλεγχο συμμόρφωσης ε, όσον αφορά αυτό το τομέα στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο εξετάζουμε και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο το γεγονό ότι άλλαξε το ρυθμιστικό πλαίσιο εν ώψη τη ε, ε κρίση και τουλάχιστον ε, τρει από τι τέσσερι ε, αρχέ εποπτεία θα αποκτήσουν και νέε αρμοδιότητε. Υπάρχει νομοθετική πρόταση της Επιτροπής ε, ε, για το ελεκτικό συνέδριο που θα, όπου το ελεκτικό συνέδριο θα ασκεί έλεγχο και υποπτία σε αυτέ τι τρει ε, εποπτικές αρχέ. Όμω αυτά αρκούν. Μήπω θα πρέπει να, να ε, έχουμε περισσότερε αρμοδιότητε για να ε, κάνουμε αυτό που κάνουμε για παράδειγμα προ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου εξετάζουμε την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τουλάχιστον να διερευνηθούν και οι δυνατότητε αυτέ. Και τέλο, υπήρξε μία ερώτηση για την απλοποίηση των δαπανών. Βεβαίω και πιστεύω και δεν χρειάζεται να σας το πω ότι ε, εγώ πιστεύω ακράδαντα σε αυτή την ιδέα της απλοποίησης των δαπανών ε, των ε, κονδυλίων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αυτό το αναφέρουμε επανειλημμένα στις ετήσιες εκθέσεις. Και αν εξετάσετε τώρα και το σχέδιο έκθεσης ε, της απαλλαγής, θα δείτε ότι αναφέρεται, αναφέρεται μίσο όπως η κοινή αγροτική πολιτική, η συνοχή και οι ιστορικές πολιτικές. Πιστεύω λοιπόν ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ε, το ζήτημα και το βλέπουμε την ίδια σκοπιά και βεβαίως πρέπει να προσέξουμε το, το ότι ε, η, η απλούστευση δεν είναι κάτι το απόλυτο Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη ετήσια έκθεση για το 2007 αναφέραμε περιπτώσεις που αφορούσαν την κοινή αγροτική πολιτική και όπου η υπερβολική απλοποίηση και απλούστευση οδήγησε σε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Εδόθη υποστήριξη από τα, ευρωπαϊκά, από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγροτικές επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα σιδηροδρομικές εταιρείες ε, ή εταιρείες γκολφ. Η κυρία Ντράσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση για τον κύριο Κίνστ. Αναφέρατε στους στόχους για το μέλλον ότι θέλετε να συνεισφέρετε στην ε, αποτελεσματικότητα στην παραγωγή εκθέσεων και συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια όσον αφορά τον έλεγχο των ε, κονδυλίων που είναι υπό κοινή διαχείριση. Αναμένεται αιτήσιε δηλώσεις από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ή θα μοιράσετε τη δουλειά μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Εθνικών. Στην κυρία Καλιουλέιτ. Δεδομένου του ότι έχει ασχοληθεί με έναν τομέα με σημαντικό ποσοστό σφάλματος μπορείτε να μας εξηγήσετε πού βρίσκονται οι υποθέσεις που έχουν αποσταλεί στον Όλαφ και να μας πείτε εάν η επιτάχυνση αποστολής υποθέσεων των Όλαφ θα αποτρέψει περαιτέρω παρατυπίες και θα επιταχύνει την ανάκτηση χρεωστήτως ε, καταβληθένων κονδυλίων. Και προς τον κύριο Λουτμπόρς αναφέρετε στόχους σας πώς ε, σκοπεύετε να βελτιώσετε την ε, δήλωση αξιοπιστίας. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα του πώς θα γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ σύντομες απαντήσεις. Σας έχετε το λόγο. Yeah. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα για την εμπλοκή των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων. Μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο πραγμάτων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας. Εμείς είμαστε υπέρ της συνεργασίας, είναι σαφές. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία των ε, τεσσάρων κρατών ε, μελών και ελεγκτικών συνεδρίων για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Όταν εξετάζαμε λεπτομερώς το εύρος ε, και την προσέγγιση του ελέγχου στα διάφορα κράτη-μέλη διαφέρει. Οπότε υπό το φως του στόχου αυτού της συνεργασίας το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκίνησε την δημιουργία αυτών των κοινών ομάδων εργασίας για κοινά ελεγκτικά πρότυπα και όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας και όσον αφορά τον έλεγχο επιδόσεων. Και η ομάδα αυτή εργασίας κοντεύει να ολοκληρώσει το έργο, το έργο της και θα πρέπει να υπάρχει ένας ενοποιημένος τρόπος ε, κοινή διαχείρισης ε, και βεβαίως ε, έχουμε και τις, τους κοινούς πιλωτικούς ελέγχους με τα επιλεγμένα αυτά ελεγκτικά συνέδρια. Μεταξύ αυτών λοιπόν που παρουσίασαν ήδη εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας επιλέξαμε τρία εθνικά ελεγκτικά συνέδρια από τη Δανία, την Τσεχία και την Ολλανδία που συμφώνησαν μαζί μας σε αυτά τα νέα πρότυπα ελέγχου. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσει κοινός έλεγχος για τα κεφάλια υποκοινή διαχείριση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βαστούν πιο πολύ ο ένας στο, ε, στη δουλειά του άλλου στο μέλλον. Και αν αυτό επεκταθεί και στα υπόλοιπα ελεγκτικά συνέδρια. Ελπίζουμε δηλαδή να γίνει αυτό με το παράδειγμα που ξεκίνησε, ελπίζουμε να επεκταθεί αυτή η συνεργασία για να βασιζόμαστε ένα στα αποτελέσματα του άλλου. κυρία Καλιουλάιντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν επανέρχονται από την αποστολή οι ελεγκτές, πολύ σύντομα γίνεται μια συνάντηση όπου συζητούνται όλα τα ευρήματα και όταν διαπιστώνεται ότι κάτι πρέπει να δοθεί στην ΟΛΑΦ, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια βεβαιότητα, το κάνουμε. Φυσικά το ταχύτερο, το καλύτερο. Ο τρόπος που λειτουργούμε επιτρέπει ε, να μειώσουμε το χρόνο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πάρα πολύ συχνά ελέγχουμε πληρωμές οι οποίες έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο και διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ε, εδώ και πάμε πολλά χρόνια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουν. Ακόμα και αν είναι σημαντικό λοιπόν τα ευρήματά μας ε, ε, να ανακοινώνονται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει την ΟΛΑΦ να προχωρά σε διαδικασίες που οδηγούν σε ανακτήσεις προγραμμάτων. Οι περισσότερες βέβαια παρεμβάσεις της ΟΛΑΦ δείχνουν ότι τα προβλήματα τα οποία σημειώνονται είναι προβλήματα παρατυπιών και λαθών περισσότερο παρά απατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης των δηλώσεων αξιοπιστίας. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Προσπαθούμε να εξετάσουμε κάθε χρόνο, κάθε δαπάνη, κάθε τομέα πολιτικό στον οποίο υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και να δούμε πώς εκτελείται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εμείς έχουμε οργανωθεί ανάλογα με τις πολιτικές τις οποίες επενδύουμε. Η πρότασή μου θα ήταν να αναδιαρθρώσουμε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, να βγάλουμε από την κοινή αγροτική πολιτική την ανάπτυξη της υπαίθρου, κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή περισσότερη, και ίσως να διευρύνουμε κάποιες άλλες πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε βάζοντας δυνατότητες πιο συγκεκριμένης μορφής ελέγχου κάποιων τομέων στο εσωτερικό των πολιτικών αυτών. Πάντως θα πρέπει σε, κάθε, σε αιτήσια βάση να ελέγχουμε τις πολιτικές τις οποίες έχουν εντοπιστεί προβλήματα στο παρελθόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, για δεύτερη φορά δεν θα θέσω ερωτήματα, εφόσον είναι η δεύτερη φορά που είστε υποψήφοι, θα κάνω μία αξιολόγηση. Έχουμε τώρα μπροστά μας τους υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Ενεκτικό Συνέδριο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω ως πρώην για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, για τα διορθωτικά ταμεία, για τον Γαλιλαίο. και μετά από τη συνεργασία με τον κύριο Κίνστ και την κυρία Καλιουλάιντ είναι το εξή. Διαπιστώνω πως ήταν πολύ συνεργάσιμοι υποψήφοι την τελευταία θητεία. Κύριε Κύριε Λιμπεράση, σα ζητώ συγγνώμη. Σε αυτή τη φάση έχουμε μόνο τι ερωτήσει. Τι αξιολογήσει θα τι κάνουμε στη συνέχεια όταν θα έχουμε τη συζήτηση και των θυρών. Αυτό ο χρόνο ε, προβλέπεται αποκλειστικά για ερωτήσει και όχι για αξιολογήσει επί των μελών. Αν έχετε ερωτήσει, ε, καλώ, διαφορετικά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Εντάξει, τότε θα, θα περιμένω και θα μιλήσω μετά στην αξιολόγηση. Ευχαριστώ, Deutsch. Ευχαριστώ. Αγαπητοί υποψήφοι. Ακούσαμε τους ε, νέους ε, υποψηφίους. Ε, όλους τα ίδια πράγματα ρωτήσαμε και θα ρωτήσω και σας τα ίδια πράγματα. Το εξής δηλαδή. Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ του ελεγκτικού συνεδρίου και του Όλαφ. Και ποια είναι η επαγγελματική σας θέση όσον αφορά την προτινόμενη θέση του Όλαφ εκτός Κομισιών και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μήπως ε, όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει και επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της απάτης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γύρω από το θέμα της σχέσης μας με την ΟΛΑΦ, το ελεγκτικό συνέδριο και η ΟΛΑΦ ε, είναι θα έλεγα καταδικασμένα όργανα σε σωστή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή ακολουθεί δύο δρόμους. Πρώτα, όταν ανοιχνεύουμε συγκεκριμένες υποθέσεις, όταν έχουμε κάποιες υποψίες ότι υπάρχει μια ποινική πράξη ή ότι υπάρχει μια απάτη, τότε προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει εγκληματική πρόθεση και παραπέμπουμε την υπόθεση στην ΟΛΑΦ. Και η ΟΛΑΦ μας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το πρόβλημα. Το δεύτερο τρόπο συνεργασίας που έχει και αυτός πολύ μεγάλη σημασία, είναι οι στενές επαφές με την ΟΛΑΦ σε επίπεδο ομάδων ε, ελέγχου και επιθεώρησης. Καλούμε στις διάφορες ομάδες τις οποίες έχουμε εμεί στο συνέδριο τους εκπροσώπους της ΟΛΑΦ και μας μεταφέρουν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους για τις προβληματικές περιοχές τους τομείς ελέγχου τους. Και έτσι προσπαθούμε να προλάβουμε ε, καταστάσεις. Ε, επίσης υπάρχουν και μόνιμα δίκτυα επικοινωνίας με την Ολάφ, στα οποία συμμετέχουν κάποιοι δικοί μας εκπρόσωποι. Σχετικά με την ε, εξωτερικοποίηση της ε, προσπάθειας της ΟΛΑΦ. Δεν ξέρω αν το συνέδριο πρέπει να παρέμβει σε αυτή τη συζήτηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι η ΟΛΑΦ προς το παρόν, σαν τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υποφέρει από έλλειψη ανεξαρτησίας. Δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γιατί να υπάρξει εξωτερικοποίηση. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί απορία, δεν είναι κάτι το οποίο απαντά στις απορίες τις οποίες έχω. Ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία, εν πάση περιπτώσει, μιας εξωτερικής ε, ε, παροχής υπηρεσία στον τομέα της ΟΛΑΦ. Από την άλλη η ΟΛΑΦ έχει συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία παρακολουθεί. Η ΟΛΑΦ ε, έχει να αντιμετωπίσει 27 διαφορετικά ε, νομικά συστήματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ΟΛΑΦ μερικές φορές ε, να μπορεί να ολοκληρώνει τις διαδικασίες αυτές με το αποτέλεσμα το οποίο κάθε φορά είναι επιθυμητό να στέλνει κάποιον εν πάση περιπτώσει στη φυλακή όταν διαπιστώνεται ένα πρόβλημα. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει πάντα. Πριν έξι χρόνια μου είχατε θέσει τις ε, ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη αυτή, ε, ε, με το συγκεκριμένο τομέα και έδωσα και την ίδια απάντηση. Απάντησα ήδη στις ερωτήσεις αυτές πριν έξι χρόνια. Είναι καλή ιδέα το να υπάρχει ένας Ευρωπαίος εισαγγελέα. η συνθήκη το προβλέπει οπότε δεν τίθεται θέμα συζήτησης να πω ότι το θέμα της ανεξαρτησίας είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και σε επίπεδο αρχής αλλά και σε επίπεδο πρακτικό. Και συμφωνώ με όσα είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, αν και το θέμα της ανεξαρτησίας, αν εξωτερικευθούν οι αποστολές της ΟΛΑΦ, ίσως να καλύψει περισσότερο τις ανησυχίες του κοινού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντμπορς, όσον αφορά την ΟΛΑΦ, συμφωνώ με τους προηγούμενους συναδέλφους δεν πιστεύω ότι δεδομένων των συνθήκων θα έχουμε εξωτερική ανάθεση της εργασίας της Όλαφ. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις και ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο και στην Όλαφ. Επειδή το ελεκτικό μας έργο πρέπει να εξετάζεται ως συμβολή, ως input στην εργασία της Όλαφ, εκτός από τις δικές τους ε, άλλες αρμοδιότητες. Όσον αφορά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ε, ε, ή την εξωτερική ανάθεση γενικότερα, δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά σημειώνω ότι ο κύριος Μπαρόζο ε, στην δεύτερη επιτροπή Μπαρόζο ανέλαβε συγκεκριμένε δεσμεύσει. Θα έλεγα ότι έχω μία σημαντική επιφύλαξη. η Όλαφ εκτός της Επιτροπής τι να σας πω, το θέμα είναι θέμα αντίληψης ε, και εικόνας της όλα εκ των έξω. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα προς αυτή την, ε, την αποθέτηση εκτός της Επιτροπής. Και όσον αφορά το γραφείο του Ευρωπαίου ε, Εισαγγελέα, σας παραπέμπω στη συνθήκη, στην συνθήκη τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και σε ένα από τα σχέδια ψηφίσματος απαλλαγή που είδα, και εσείς αναφέρεστε ε, στο ότι θα πρέπει να υπάρξει η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με το πόσο σύντομα θα δημιουργηθεί. Ο, κύριο ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας ε, κατά τη διάρκεια τη εντολή σα. Να πω στον κύριο Λούτσπορκ... ο οποίο μα είπε ότι υπάρχουν 20 κενέ θέσει ελεγκτών. Και εγώ προσκρούω στο πρόβλημα αυτό. Συχνά ε, το τονίζουμε. Μην διστάζετε να επικοινωνείτε με, τους, ε, με, τους, ε, με τα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί εδώ είναι ζήτημα. Δεν μπορεί να συζητάμε συγκεκριμένε εργασίε και να μην έχετε τα μέσα. Τώρα, πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσει. Όσον αφορά το, χρονο, το χρονοδιάγραμμα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα δώσει όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά. Ε, μέχρι την 21η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου μπορούμε να έχουμε ε, την έκθεσή σας για το έτος που ακολουθεί ε, το, το ελεγχόμενο οικονομικό έτος, γιατί πραγματικά η διαδικασία απαλλαγής παίρνει πολύ χρόνο. Και εσείς δεν μπορεί... Κοίτα, κάνετε κάποιες παρατηρήσεις στην έκθεσή σας, αλλά τόσο όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, το ελεκτικό συνέδριο έδωσε γνωμοδότηση, αλλά δεν ε, έδωσε το πράσινο φως, δεν μίλησε για την αξιοπιστία ε, των ενεξελίξη ε, συναλλαγών. για τη τελευταία ανάλυση δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον ΤΑΣ. Από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχουμε συνολικά ΤΑΣ, συνολικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Ευχαριστούμε. Κύριος Κίνστ. Yes, uh, Όσον αφορά αυτό το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι ανοιχτό να συζητήσουμε αυτές τις ε, δυνατότητες αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Αλλά με την εξαετή μου εμπειρία, κυρίως στον τομέα ε, των τάς, των δηλώσεων αξιοπιστίας, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτή την ε, ε, σύντμηση των διαστημάτων. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος του ελέγχου, του, της ε, του ελέγχου και της γνωμοδότησής μας. Δηλαδή, κοιτάξτε, για τη γνωμοδοληψία, για παράδειγμα, πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους ε, κανόνες και τα τελευταία δείγματα των συναλλαγών που αποτελούν το αντικείμενο ελέγχου θα πρέπει να, γίνονται, να, να λαμβάνονται από τι ε, συναλλαγέ που γίνονται στο τέλος του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη. Στη δική μου την περίπτωση εδώ μιλάμε και για χώρε ε, που βρίσκονται στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τι εσωτερικέ διατάξει, διαδικασίε ελέγχου. Ε, και μερικέ φορές ε, στη διαδικασία καθάρισης η Επιτροπή μα διορθώνει. Όταν αξιολογούμε κάτι ως φάλμα και στη συνέχεια βλέπουμε τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ε, αποδεικνύουν το αντίθετο, διορθώνουμε κτλ. Μέσα Νοέμβρη λοιπόν ε, εκεί μπορούμε να είμαστε ε, ε, σίγουροι ότι όταν λέμε 11% σφάλμα στα διαφορετικά ταμεία, αυτό το 11% είναι σωστό. Άρα, σας λέω ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι ανοιχτό και μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά μετά από την εμπειρία που έχω και εγώ στα έξι χρόνια, νομίζω ότι όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου από μεριά ελεκτικού συνεδρίου, τα περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά. Δεν ξέρω, μπορώ να συνεχίσω με τις άλλες ερωτήσεις. Μάλιστα. Ο κ. Ναι, έχετε δίκιο. Οι προσεγγίσει είναι, δύο διαφορετικές, είναι και οι απόψεις είναι διαφορετικές ανάλογα με τους λογαριασμούς. Έχουμε μία γνωμοδότηση για την αξιοπιστία των λογαριασμών και όσον αφορά την νομιμότητα ε, και την έλλειψη παρατυπίας ε, των βασικών συναλλαγών, εδώ έχουμε μικρότερες ε, ε, δηλώσεις αξιοπιστίας, ε, υποδηλώσεις για κάθε τομέα. Κατά την άποψή μου το σύστημα αυτό είναι διαφανέστερο, γιατί κοιτάξτε, ε, είναι μοναδικό στη φύση του ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει διαφορετική φύσεω δαπάνε, διαχείριση και κινδύνου. Ίσως λοιπόν εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου θα βλέπατε ότι η διαδικασία είναι λιγότερο διαφανής εάν είχαμε μία και μόνο DAS για όλες τις συναλλαγές αναμειγνύοντας τα διευθυντικά ταμεία, ε, τις διοικητικές δαπάνες, την εκπαίδευση, εξωτερική δράση κτλ. Άρα, όπως σας είπα, στόχος μας είναι να είμαστε στις νομοθετήσεις μας ώστε με τον πιο διαφανείς για, τις, ε, ε, για τους διάφορους τομείς δαπανών. Ίσως βέβαια θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε κατά πόσον αυτές οι ομάδες δαπανών που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου αυτή τη στιγμή ε, χαρακτηρίζονται από την κατάλληλη ισορροπία ή κατά πόσον θα πρέπει να κάνουμε μια αναδιάρθρωση. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν καλή ιδέα να έχουμε μια συνολική DAS. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σας ευχαριστώ. Thank you, Κύριε Κατζουλάιτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά τη συνοχή, να σα δώσω ορισμένε ημερομηνίε. Οι τελευταίε συναλλαγέ, οι τελευταίε παρατυπίες συναλλαγέ, Μάλλον, ε, οι τελευταίες συναλλαγές είναι ορατές στις 15 Ιανουαρίου ε, και οι τελευταίες ε, δαπάνες πάνω από το 11ο καταλαβαίνετε ότι γίνεται στο τέλος του χρόνου. Υπάρχει αυτή η βιασύνη προς το τέλος του χρόνου. Και πραγματικά πρέπει να δούμε εκεί τι γίνεται σε αυτές τις πληρωμές που γίνεται το Δεκέμβρη. Δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Εάν ε, κάνουμε νωρίτερα τη δειγματοληψία, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. 15 Ιανουαρίου έχουμε δειγματοληψία από τις τελευταίες πληρωμές χρειάζονται, ε, απαιτούνται και έξι εβδομάδες ε, για να συμφωνήσει το ε, κράτος μέλος. Είμαστε έτοιμοι μέσα Φεβρουαρίου. Ο έλεγχος παίρνει τρει εβδομάδες. Ωραία, εδώ μπορούμε τις τρει εβδομάδες να τις κάνουμε δύο εβδομάδες και να υποβάλουμε έκθεση σε δύο εβδομάδες. Πάμε μέσα Μαρτίου. Το κράτος μέλος έχει 8 εβδομάδες να απαντήσει. Άρα ήδη φτάσαμε στο Μάιο. Και μόνο τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το τριμερές σύστημα το οποίο έχουμε θεσπίσει. Αν λοιπόν ε, πιέσουμε ιδιαίτερα τι ημερομηνίε, φοβάμαι ότι πάλι θα καταλήξουμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πριν από λίγα χρόνια, όπου είχαμε ε, αντιφατικέ διαδικασίε και εδώ στην ε, Σακροάση Κοκομπού. Βεβαίω, κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο. αυτό σημαίνει ότι οι προθεσμίε θα πρέπει να ε, συντμηθούν για όλου. Αλλά όλε οι τεχνικέ διαδικασίε και η μετάφραση που δεν είναι αμεληταίο πρόβλημα καταδεικνύουν ότι μάλλον δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίση, τα ποσοστά ασφάλματο που υποβάλλουν ε, τα κράτη-μέλη στον τομέα τη συνοχή φτάνουν το Δεκέμβριο ε, συνένα, δηλαδή του επόμενου έτου. σω λοιπόν αυτά θα μπορούσαμε να τα λάβουμε υπόψη, ε, θα λάβετε υπόψη όταν ξεκινάτε τη συζήτηση για την απαλλαγή. Αν όλη η συζήτηση γίνει νωρίτερα, ε, τότε και, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και εδώ το, το, το, την πτυχή ελέγχου. Δεν είναι κάτι λοιπόν που λύνεται μέσα σε μία μέρα. Απαιτείται μια, πολύ, ε, ε, ομάδα εργασία που να εργαστεί εντατικά, αν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Συνολική, μια τάση, συνολική τάση. Ίσως σε κάποιο σημείο, όταν τα ποσοστά σφάλματος είναι ε, χαμηλά παντού σε όλα τα σημεία του προπολογισμού, εκεί θα πρέπει να δούμε κατά πόσα θα μπορούσαμε ε, να έχουμε μια θετική αρνητική τάση, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι συναλλαγέ και τι υποκείμενε. Αν φτάσουμε όμω σε χαμηλό επίπεδο σφαλμάτων σε όλου του τομεί. Τώρα όμω, όπου ορισμένε ε, εκθέσει αξιολόγηση παρουσιάζουν πολύ σημαντικό ποσοστό σφάλματο, δεν ξέρω πώ μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Και να μην ακολουθήσουμε την οδό των ειδικών αξιολογήσεων. Γιατί καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εάν, όπως σας είπα, ε, αλλάξουν τα πράγματα, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι όσον αφορά την ε, παρατηρήσή σας για τις θέσεις που αναζητούμε πράγματι θα μας βοηθήσει η στήριξη του Κοινοβουλίου όπως ξέρετε για τον προβολισμό του 2011 υπάρχει μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών και οπωσδήποτε θα μας βοηθούσε να αποκτήσουμε τις θέσεις τις οποίες ε, θέλουμε τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας ε, για το να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας το συντομότερο δυνατόν, αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι και κατά την άποψή μου η ταχύτητα είναι εις βάρος ποιότητας. Μπορεί να γίνει γρήγορα, αλλά δεν ναι, θα είναι τόσο υψηλή ποιότητα. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Μήπως είναι καλύτερο να έχουμε χρόνο να κάνουμε τη δουλειά μας ε, σωστά. Και αντί για Νοέμβριο, δηλαδή τώρα αντί για Νοέμβριο να βγάλουμε την έκθεση Οκτώβριο, δεν ξέρω κατά πόσον όφελη και κατά πόσο είναι εφικτό να έχουμε την ίδια ποιότητα που έχουμε τώρα. Για την τελευταία σας ερώτηση για την συνολική δήλωση αξιοπιστίας πράγματι έχετε δίκιο. Πράγματι, πως ε, δεν υπάρχει μια γενική δήλωση αξιοπιστίας. Κατά την άποψή μου, ε, καλό είναι να μην ανακατεύουμε διαφορετικά πράγματα και να τα βάλουμε όλα μαζί και να, πούμε, να βγάλουμε συμπεράσματα συνολικά για πράγματα που είναι διαφορετικά και από τη φύση τους και από τη διαχείρισή τους και θεωρώ πως ε, το τρέχον σύστημα που κάνουμε εξχωριστή αξιολόγηση είναι αρκετά καλό. Βεβαίω, μπορούμε μετά να δούμε πώς ε, μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο οι εθνικές δηλώσεις ε, που θα έχουν ελεγχθεί με τα πρότυπα του ελεγκτικού συνεδρίου. Εάν ναι, συμβεί κάτι τέτοιο νομίζω καλό θα είναι τότε να επανεξετάσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σοντή πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πια χρόνο. θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία λέγει η συνθήκη. Η συνθήκη ζητά από το ελεγκτικό συνέδριο να δώσει δύο διαβεβαιώσεις. Τη μία σχετικά με τους λογαριασμούς και τη δεύτερη τη σχετική με τις συναλλαγές. Και μπορεί να κάνει παρατηρήσεις σε τομείς δραστηριότητας, κάτι το οποίο το κάνετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο δεν κάνετε αν θέλετε είναι η γνωμοδότηση για τις συναλλαγές. Αυτό δεν είναι μια πολιτική φιλοδοξία την οποία έχουμε. Καλώς, ευχαριστώ, δεν έχουμε πλέον χρόνο. θα πρέπει να προχωρήσουμε και κλεισμένων των θυρών από εδώ και πέρα στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων των υποψηφίων.